Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ως ήθιστε, θα αρχίσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Είναι πολύ σημαντικό. Αύριο, 5η, 22 Μαρτίου, 9 με 12.30, να ξέρετε ότι δεν θα λάβει χώρα συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και αυτό γιατί Φύγαν από την ημερήσια διάταξη κάποια σημεία που είχαμε προβλέψει για αύριο. Οπότε δεν θα υπάρξει η αυριανή συνεδρίαση καθόλου. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται. Σύμφωνοι. Ωραία. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν έχω. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 22 και 23 Ιανουαρίου 2018. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις επί των πρακτικών αυτών μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και ερχόμαστε στο πρώτο ουσιώδες θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα, το σημείο 4. Πρόκειται για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα Ίσως έχουμε καθυστερήσει λίγα χρόνια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει παραμένει πολύ επίκαιρο. Πρόκειται για την εξέταση ερώτηση με έτοιμα προφορική απάντηση και ο εισηγητή μας είναι ο συνάδελφος Μάρκος Πίπερ. Έχουμε και τους σκιώδει εισηγητέ, ε, βέβαια. Ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των mid-caps είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει οριζόντια διάφορους τύπους νομοθεσίας. Εμείς στην Επιτροπή μας Ήτρε είμαστε υπεύθυνοι για το Κόσμε που είναι ένα πολύ ειδικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την καινοτομία. Η προφορική ερώτηση της ΙΤΡΕ, λοιπόν, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει, σκοπεύει να προωθήσει την διευκρίνηση του ορισμού αυτού και την επανεξέτασή του, προκειμένου να υπάρχει ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο και πιο δίκαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις mid-caps. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι διαθέτουμε 45 λεπτά για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση δηλαδή πριν τις 10. Λοιπόν, για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, θέλω ο εισηγητής, ο συνάδελφος κ. Πίπερ, να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Μάρκος, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν ώρα να συσχοληθούμε το θέμα αυτό. Αυτή η προφορική ερώτηση γίνεται στα πλαίσια ακριβώς της διαδικασίας διαβούλευσης που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορά το ότι δεν έχουμε κανέναν ορισμό για το τι σημαίνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ μεταξύ μας τώρα δεν χρειάζεται να σας περιγράψω αναλυτικά τη σημασία των μικρομεσαίων. Ξέρουμε ότι είναι περίπου 25 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσει στην Ένωση με βάση τον ορισμό που έχουμε τώρα. Και ίσως να εκπλήξει πολλούς το εξή. 75% ενός γιοταχή παράγονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι από μεγάλα, μεγάλους ομίλους. Βεβαίως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι βαθιά ριζωμένες στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης και έχουν ε, τη διασύνδεσή τους ε, με πολλές άλλες επιχειρήσεις στην ίδια περιφέρεια, άρα συμβάλλουν ιδιαίτερα στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας. Οι μικρές επιχειρήσεις φυσικά επηρεάζονται, όπως και συνολικά οικονομία, από το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ευρεία διακομματική συνένεση ότι μια επιχείρηση που δεν έχει μεγάλο διοικητικό τμήμα, δεν είναι δυνατόν να έχει τόσο πολλές υποχρεώσεις είτε για την προστασία των δεδομένων, είτε για το τι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται, είτε για πολλά άλλα θέματα. Όλες αυτές οι προδιαγραφές οι νομοθετικές, ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις ε, τις φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχουν όλους αυτούς τους ειδικού για να ασχοληθούν με όλα τα θέματα αυτά. Δεν έχουν ούτε τους πόρους για να έχουν έναν επιφορτισμένο με την προστασία των δεδομένων, έναν ειδικό για την ε, επιτήρηση των συνθήκων εργασίας δεν έχουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ε, γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τη δική μας πολιτική, πώς να υποβάλουν αιτήσει, για παράδειγμα για να παίρνουν επιδοτήσεις με επιτυχία. Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτός ο ορισμός των μικρομεσαίων, όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η ανισότητα και η άνηση μεταχείριση είναι των μεγάλων και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Για παράδειγμα για την πρόσβαση στο κόσμο, στο ορίζον 2020, ε, στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να υπάρχουν κάποιες ποσοστός για τις μικρομεσαίες και να υπάρχει και μια ελάφρυνση της γραφειοκρατίας για την υποβολή των αιτήσεων. Αλλά και σε άλλους τομείς, ως Ευρωπαίοι νομοθέτες, έχουμε επιτρέψει εξαιρέσεις. Για παράδειγμα για το εμπόριο των πιστοποιητικών ε, ε, για τις εκπομπές αερίων. Βεβαίως ε, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες για τις εκπομπές, αλλά υπάρχει μια ελάφρυνση της γραφειοκρατίας. Γιατί τώρα ξαναπροσπαθούμε να ασχοληθούμε με τον ορισμό των μικρομεσαίων. Έχουμε έναν που ισχύει εδώ και καμιά 15 ετία. Αλλά εντωμεταξύ βεβαίως έχουν υπάρξει εξελίξεις, οπότε θεωρώ ότι αναγνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να βασιζόμεθα μόνο στην, στον αριθμό των απασχολουμένων και στον κύκλο εργασιών. Πρέπει ε, να υπάρξει μια αναπροσαρμογή των ορισμών. Σε τι βαθμό και σε σχέση με την υψηλότερη παραγωγικότητα ε, πρέπει να το συζητήσουμε βέβαια. Αυτή είναι η πρώτη προσαρμογή που προτείνουμε. Η δεύτερη πρόταση που κάνουμε είναι αλλά οι επιχειρήσεις επίσης προτείνουμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις ε, που δεν ανήκουν πλέον στις μικρομεσαίες γιατί έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους θα πρέπει να έχουν μια περίοδο προσαρμογής, μια μεταβατική περίοδο. Τρίτον, βεβαίως ξέρουμε ότι ορισμένοι ε, μεταχειρίζονται με λάθος τρόπο αυτό τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταχρώνται αυτών των δυνατοτήτων που τους δίνουμε. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να φροντίσει να μην υπάρχουν περιθώρια καταχρήσεων. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε σωστά τους στόχους για να βοηθάμε τις σωστές μικρομεσαίες, τις πραγματικές μικρομεσαίες. Επίσης πρέπει να απομακρυνθούμε κάπως από τα καθαρά ποσοτικά κριτήρια, αριθμός εργαζομένων, κύκλος εργασιών και να οδεύσουμε προς κριτήρια που να είναι πιο ουσιώδη. Για παράδειγμα, αν οικογενειακή επιχείρηση, αν εξάγει πολλά, αν υπάρχει υψηλή παραγωγικότητα, πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις, ούτω ώστε να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση στο διεθνές εμπόριο. Για παράδειγμα, ήδη μέσω του ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ήδη μέσω του ΕΦΣΥ, έχουμε τον ορισμό των μικρών εταιριών μέσης κεφαλαιοποίησης small mid caps. Και αν δούμε για παράδειγμα τις νέες πρωτοβουλίες μέσω του Ταμείου Άμυνας, υπάρχει δυνατότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μέχρι 3.000 εργαζομένους για το Ταμείο αυτό. Πρέπει λοιπόν να απομακρυνθούμε από τα ποσοτικά προς ποιοτικά κριτήρια. Δηλαδή, ο στόχος Δεν θέλουμε να δυσχεράνουμε την κατάσταση για τις επιχειρήσεις που είναι, που είναι ήδη σε αυτόν τον ορισμό. Όχι. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλες τις επιχειρήσεις για απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Θέλουμε να υπάρχουν περισσότερο ποιοτικά κριτήρια. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας, για την παρουσία σας. Η κυρία Πατρίτσια Τόια είναι σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους των ε, σοσιαλιστών και πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήτρε. έτσι. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πω προς τον συνάδελφο ότι εκτιμώ τις προθέσεις του και τον απότερο, τους απότερους στόχους του, αλλά θα πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι έχω πολλαπλές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, ιδιαίτερα ως προς την πρόταση ψηφίσματος, όχι την προφορική ερώτηση και είναι αντιρρήσεις γιατί κατά την άποψή μου αυτή η πρόταση ψηφίσματος είναι αντιφατική γιατί αντιμετωπίζει τον θέμα των ΜΜΕ πέρα από τις ε, διαστάσεις στα κράτη-μέλη γιατί ε, υπάρχει ένας ορισμός ε, σε σχέση με το μέγεθος παρά τις διαφορές. Τώρα, το να συγχέουμε το θέμα των ΜΜΕ με τις εταιρείες ε, μεσαίας κεφαλαιοποίησης ε, είναι οξύμορο και στην ουσία διαστρεβλώνει τις ΜΜΕ, τον ορισμό των ΜΜΕ, διότι μιλάμε για ένα 1% όταν μιλάμε για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ανισότητα, γιατί έχει σημασία το πώς θα υποστηρίξουμε και φορολογικά της ΜΜΕ στην πλειονότητα των κρατών μελών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αντιφατικό αλλά και επικίνδυνο ε, κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για ΜΜΕ ή για ΜΚΑΠΣ. Έχει μεγάλη διαφορά. Επίσης, στις ΜΜΕ θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα εξαγωγών ως κριτήριο. Δηλαδή, προβάλλουμε κυρώσεις κατά των ΜΜΕ που δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν στις αγορές, να προβούν σε εξαγωγές. Γι' αυτό δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με τις ε, εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επίσης, Μιλάμε για μια βιομηχανική πραγματικότητα η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μεγέθη. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λήξει, νομίζω ότι θα λήξουν κατά τα μέσα Μαΐου. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε την πρόταση ψηφίσματος. Άρδιν, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με τον ορισμό των ΜΜΕ. Thank you uh, very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ τώρα, ο κύριος Μπασίρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προέρχομαι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκλέγομαι βουλευτής έχοντας δουλεύει 35 χρόνια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, χαίρομαι που η Επιτροπή μας δημιούργησε αυτή την ομάδα και προσπαθεί να καταλήξει σε έναν ορισμό για το ποιε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις στηρίξει. Πράγματι, προσφέρουν ε, πάρα πολύ απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς κάθε βοήθεια που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι θετική για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με την ομοθεσία και την γραφειοκρατία καλύτερα. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι ευπρόσδεκτοι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές στο έργο τους και να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην ουσία του έργου τους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Πίπερ, τον εισηγητή, για το ψήφισμα που ετοίμασε όσον αφορά τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο κειμένου λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τη σήμερα ημέρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όπως είπα και νωρίτερα, το διοικητικό άχθος, για παράδειγμα, που τους επιβάλλεται. Συχνά ε, μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νομοθετικά κείμενα. Τώρα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα πόσο ζωτική σημασία είναι για την οικονομία μας. Και προσβλέπω και εγώ στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε για τις παρατηρήσεις σας. Επόμενος ομιλητής τώρα, εκ μέρου τη Άλτερ, η κυρία Νέκτιγκαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Πίπερ για το έργο του. Όμως ειλικρινά εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ τη χρήση αυτού του ορισμού που προτείνεται. Και θα ήθελα να προτείνω τροπολογίες σε αυτά που ζητάει το ψήφισμά μας. Για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι ο ορισμός δεν θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο. Αντίθετα, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει την εφαρμογή που έχουμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω και κάποιες ανησυχίες για το γεγονός ότι αναφέρεται ο αριθμός των εργαζόμενων και ότι δεν θα έπρεπε να αποτελέσει κριτήριο εφ' για να δούμε κατά πόσο μια επιχείρηση είναι ή δεν είναι μικρόμεσα επιχείρηση. Γιατί όχι. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έχουμε δουλέψει με το κριτήριο αυτό του αριθμού των εργαζόμενων, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια. 15 χρόνια και είναι ένα αποδεκτό κριτήριο αυτή τη στιγμή παντού στην Ευρώπη για 99% όλων των επιχειρήσεων. Οπότε θέλουμε να υποβάλουμε τροπολογίες από αυτού. Και όπως είπε και ο προλαλής σας, και εμείς προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ, η κυρία Λόπες Μπελμέα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για την Ευρώπη. οικονομική σημασία, δημιουργούν πλούτο, απασχόληση. Γνωρίζουμε επίσης επαρκώς πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα και χρησιμοποιούν ακόμα τα κενά στην ομοθεσία και την πολυπλοκότητα επίσης ε, στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να παρακάμψουν τους κανόνες είτε του Ευρωπαϊκού είτε τους εθνικούς. Προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φορολογικές και εργασιακές τους υποχρεώσεις και να πάρουν ενισχύσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν. Οπότε, σωστός ο προσανατολισμός, αλλά δεν νομίζω ότι λύνεται σωστά το ζήτημα. Ε, διατυπώνεται το πρόβλημα, αλλά έτσι ανοίγει η πόρτα σε καταχρήσεις πάνω στην νομοθεσία. Και χωρίς να το θέλουμε, κατά πάσα πιθανότητα, πλήττουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάνω από το 90% δηλαδή του παραγωγικού ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός των εργαζόμενων, οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να παραμείνουν ε, κεντρική σημασία στον καθορισμό και στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι νέα στοιχεία για σχέσεις ε, επιχειρησιακές που πλήττουν τις πραγματικές μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις πρέπει να εξεταστούν πολύ περισσότερο και δεν πιστεύουμε ότι, πρέπει, ότι θα οδηγήσει κάτι τέτοιο σε περισσότερη ευελιξία. Είμαστε κατά επίσης της διεύρυνσης του ορισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν και μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα οι mid-caps βασίας ε, κεφαλοποίησης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να περιοριστούμε στις πραγματικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και σας για τις παρατηρήσεις σας. Επόμενος ομιλητής, Τάριο Ταμπουράνο από το Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ δέχομαι αυτά που είπαν οι προλαλήσοντες και πιστεύω ότι οι ΜΜΕ ε, εκπροσωπούν το 100% των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό η σύσταση του 2003 οδήγησε σε μια ιερή ισορροπία την οποία πρέπει να υπερασπιστούμε. Βεβαίως από τότε δεν έχει επικαιροποιηθεί το έγγραφο το 6, 9 ή 12 και έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις με ένα θετικό πλαίσιο ως προς το κύρος αυτού του εγγράφου και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης. Θα αρκεστώ σε αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε το σχέδιο του κυρίου Πίπερ πριν σταθμίσουμε τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία. Θα πρέπει να μην γίνει μια γενικότερη αποτίμηση. Η Επιτροπή έκανε μία μελέτη αντικτύπου σε σχέση με την αύξηση πληθωρισμού και παραγωγικότητας μέσα στα πλαίσια της κρίσης που δεν λαμβάνει υπόψη ο κύριος Πίπερ. Αυτό δεν αμφισβητεί κανένα από τα κριτήρια που ορίσαμε. Ούτε γίνεται λόγος για νέα κριτήρια όπως τον όγκο εξαγωγών και τις διάφορες δασμολογήσεις. Και ούτε προτείνεται ένας νέος ad hoc ορισμός για τις ΜΜΕ. Νομίζω ότι κατά τις διαπραγματεύσεις θα δούμε πώς θα έχουν οι εξελίξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική. Γιατί να υπάρχει προθεσμία στην 26η Μαρτίου ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Αυτό είναι πολύ ε, μικρό χρονικό διάστημα και δεν ε, το διέπει και καμία λογική. Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να μιλήσει για τις συστάσεις και για τον ορισμό των ΜΜΕ ή τυχόν τροποποίησης και με βάση αυτή την συλλογιστική δεν βλέπω γιατί να μην τηρήσουμε αυτό το πλαίσιο διαβούλευσης. Γι' αυτό ως ομάδα, η FTD, θα ήθελα η προθεσμία να τεθεί δύο εβδομάδες μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Μπένσεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των ΜΜΕ και του μεγέθους τους, όπως ε, προείπαν και πολλοί συνάδελφοι. Γιατί το 95% είναι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για τον ορισμό και να ξαναδούμε τα κριτήριά μας. Νομίζω, και εδώ εκφράζομαι προσωπικά, ε, ως πρόεδρος των ΜΜΕ Europe, των ΜΜΕ της Ευρώπης ε, και να πω ότι ζητήσαμε μία επαναξιολόγηση του ορισμού των ΜΜΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι η μεγάλη παίκτες ή επιχειρήσεις να μην δημιουργήσουν ειδικέ δομές ε, για τις ΜΜΕ για δική τους χρήση και προτέρημα. Μας ενδιαφέρουν βεβαίως και οι εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης και νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα κριτήρια που είχαμε. Γιατί θεωρούμε ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να τύχουν τις υποστήριξεις που έχουν. Γιατί οι ΜΜΕ δημιουργούν το 80% της απασχόλησης στην Ευρώπη. Άρα οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποστηριχτούν με βάση αυτό το πλαίσιο υποστήριξης της ΜΜΕ. Άρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ και όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο συνάδελφος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό θέμα ζωτικής σημασίας γιατί από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τα δύο τρίτα των ε, εργαζομένων στην Ευρώπη εργάζονται σε μικρομεσαίες. Και το 50% του ΑΕΠ μας παράγεται από αυτές τις επιχειρήσεις. Και είναι πολύ σημαντικές ε, για την εγκύτητα που έχουν προς τους πελάτες τους, τους συμπολίτες μας. Άρα πρέπει να υπάρξει απλούστευση της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε αυτή τη μελέτη για τις πιο επιβαρυντικές, τις πιο γραφειοκρατικές νομοθετικές πράξεις της Από εκεί έχουμε τις περισσότερες διαμαρτυρίες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε τώρα έναν κανονισμό για τις ε, στατιστικές, επί το οποίο θα ψηφίσουμε, που επιβάλλει και νέο διοικητικό άχθο για τις μικρομεσαίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στις μικρομεσαίες να ασχολούνται με τα προϊόντα τους και με τους πελάτες τους. Small is beautiful. Το μικρό είναι όμορφο. Έτσι λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Και για την κοινωνία ο ανταγωνισμός είναι η μόνη οδός προς την ευημερία. Και ο στόχος μας πρέπει να είναι η ευημερία. Άρα είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αυτές οι μόνο απευθυντικές θηρίδες, τα one-stop shop για τις μικρομεσαίες. Θα ήθελα λοιπόν να μην δημιουργήσουμε νέους φραγμούς, διότι είναι ήδη αρκετά δύσκολο για έναν ε, ελεύθερο επαγγελματία να προσλάβει ένα συνεργάτη. Ξέρουμε πόσο υπεύθυνο είναι αυτό. Κάθε επιπλέον εμπόδιο για οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε έχει 250, είτε 500, είτε περισσότερους εργαζόμενους, όλα αυτά θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνουν χωρίς εμπόδια. Δεν είναι δυνατό να μην μπορεί να προσληφθεί κάποιος γιατί δεν μπορεί να υπαχθεί στο α ή στο β καθεστώς εργαζομένου. Πρέπει λοιπόν επιπλέον να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν ε, όταν έχουμε τόσο, μεγάλες, τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, 22 ε, εκατομμύρια να θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε κανονισμούς που να ισχύουν ακριβώς για την κάθε μία επιχείρηση. Πρέπει να βρούμε νέες στρατηγικές που να βοηθήσουν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις αυτές να ξεκινήσουν τι εξαγωγές τους. Ευχαριστώ πολύ, Πάουλ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ο κύριος Ηλικιώτης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκαλιά της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, και των νεοφιλεύθερων μνημονιακών πολιτικών που επιβλήθηκαν, πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει αναγκάστηκαν να κλείσουν οδηγώντα στην αγία χιλιάδε οικογένειε. Να πω ότι, για παράδειγμα, στην Κύπρο, όπου οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων, δυστυχώ λόγω των πολιτικών λιτότητα και μη επαρκού στήριξη, άνω των 15.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναγκάστηκαν να κλείσουν. Είναι γι' αυτό που θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματική ε, ε για τα μικρά κράτη-μέλη την αλλαγή του ορισμού, το άνοιγμα του ορισμού και κατά την άποψή μα θα πληγούν περαιτέρω η μεγάλη πλουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να τα γνωρούμε όταν συζητάμε οποιαδήποτε, οτιδήποτε αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πόσο μάλλον όταν επιχειρείται η αλλαγή του ορισμού, το τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Για την ομάδα μα, την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, όπω ανάφερε και η συνάδελφο Παλώμα Λόπε, οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει ορισμό προκειμένου να διευρυνθεί και να καλύπτει και μεγάλε επιχειρήσει σε βάρο αυτών που είναι πραγματικά μικρομεσαίε, μα βρίσκει κάθετα αντίθετο. Έχουμε χρέο να στηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ώστε να τονωθεί η πραγματική οικονομία και να προστατευτούν χιλιάδε θέσει εργασία. Αντί λοιπόν να επιχειρείται μείωση τη βοήθεια που τη χάνουν, ζητάμε να δοθούν νέα κίνητρα ανάπτυξη, να ενισχυθεί η οικονομική στήριξη από, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθούν μέτρα για διευκόλυνση τη πρόσβασή του στη χρηματοδότηση ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ιδιαίτερη έμφαση και ειδική στήριξη των πρέπει, πρέπει να δοθεί στι μικρό-μεσαίε επιχειρήσει, στι ε, micro SMEs, οι οποίε ε, κατά κανόνα είναι οικογενειακέ επιχειρήσει και οι οποίε αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα ε, προβλήματα σε πολλά κρατημέλη και ιδιαίτερα στα μικρά κρατημέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο κύριος Εντουάρ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Με εκπλήσει λίγο αυτό που άκουσα από τον κύριο Πίπερ, ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τους 3.000 υπαλλήλους στη Γαλλία. Έχουμε ένα δίκτυο τέτοιων επιχειρήσεων με 3.400.000 ε, επιχειρήσεις και το 90% είναι κάτω από 10 υπαλλήλους. 5% έχουν 10 με 500 υπαλλήλους. Πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά όσον αφορά τον ορισμό αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποιο είναι το μέγεθος υπαλλήλων μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και νομίζω ότι όλοι ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ότι χρειάζεται ευελιξία είναι ένας παραγωγικός ιστός ο οποίος ε, πράγματι ε, μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις. Βέβαια πέρασε από κρίση ε, ο κλάδος. Οι πρώτες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονομική κρίση ήταν βέβαια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε κατά τη γνώμη μου το καθοριστικό εκεί που πρέπει να επικεντρώσουμε τον προβληματισμό μας είναι το πώς θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γιατί δεν ξέρω στις άλλες χώρες, φαντάζομαι το ίδιο γίνεται, είναι πραγματικά φοβερά δύσκολο, είναι γολγοθάς για να καταφέρει να φτάσει κάποιος στη χρηματοδότηση. Και οι τράπεζες έχουν ρόλο για να στηρίξουν την δραστηριότητα αυτού του οικονομικού κλάδου που είναι αναγκαία. Γι' αυτό και θα ήθελα έναν ορισμό αρκετά ρεαλιστικό για το τι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά συγχρόνω να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει αυτέ, ε, ποιο το επίπεδο και νομίζω, προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τελικά ο κόσμος το ε, χρηματοπιστωτικό να μπορέσει να τη στηρίξει. Είναι ζωτική σημασία για την οικονομία μα. Το είπαμε, 90% θέσεων απασχόληση προέρχονται από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω κι εγώ τρία πράγματα. Τίποτα καινούριο, όπως λέτε και εσείς συνάδελφοι, έτσι και εγώ θέλω να μιλήσω για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θέλω να αναφέρω δύο προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το COSME, πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες καινούργιες ιδέες ε, στο Συμβούλιο καινοτομία για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα έπρεπε λοιπόν να ελέγξουμε ποια είναι η μορφή του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το COSME είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για όλες τις μικρομεσαίες στην Ευρώπη. εκατό εκατομμύρια άνθρωποι που εμπλέκονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εποφελούνται από τη χρηματοδότηση του κόσμου. Η ιδέα της καινοτομίας είναι η βάση του κόσμου. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, χρηματοδότηση θέμα δηλαδή, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι 20-30% των ε, συνολικών επενδύσεων πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, όλα συμφωνούν μεταξύ τους οι προτάσεις σας, ναι, δεν λέω, όλα. είναι απαραίτητο να δούμε τι γίνεται και με το Ταμείο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Και θα πρόσθετα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να συζητήσουμε με την κοινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. φαντάζομαι και ο συγητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εμπειρία από τέτοιες ε, συζητήσεις με τον κλάδο. Μα αναφέρθηκε κιόλα. Στην αρχική σας ε, παρουσίαση, Μάρκος, το είπατε. Αλλά ε, μπορείτε να προσθέσετε κάτι. Οι οργανώσεις των μικρομεσών επιχειρήσεων είναι ισχυρές. Οπότε θα μπορούσατε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες και από αυτού θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας. Στηρίζεται τις γενικές ιδέες του ορισμού. Τώρα, ο κύριος Αντρόπουλος από τη Γενική Διεύθυνση Grow, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τα έργο της για μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όντως εντοπίζεται τα βασικά στοιχεία της συζήτησης. Πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την τροποποίηση του ορισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε στα μέσα του δρόμου ουσιαστικά. Και θα σας εξηγήσω ποιον το υπόβαθρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε τα διάφορα επίπεδα του ορισμού καθετόσο και καθετόσο κάνουμε αξιολογήσεις. Και όλες οι αξιολογήσεις μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι τέλειος, μεν, αλλά λειτουργεί καλά για τις περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, άμα συγκρίνουμε με αντίστοιχους ορισμούς σε άλλες περιοχές του κόσμου, είναι πιο κατάλληλος ο δικός μας ορισμός για τους στόχους που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 υπήρξε δικαστική απόφαση όσον αφορά μια δικητική απόφαση της ΕΚΑ που είχε να κάνει με το κατά πόσο δύο επιχειρήσεις ήταν ή δεν ήταν μικρομεσαίες. Ανέλησε λοιπόν την διοικητική αυτή απόφαση το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η απόφαση ήταν πιο περιοριστικός από ό,τι προέβλεπε ο ίδιος ορισμός. Κάτι το οποίο οδήγησε στη συνέχεια και εμείς να δουλέψουμε παραπάνω πάνω στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τι έχουμε κάνει προς το παρόν. Πρώτον, έχουμε δημοσιεύσει μια πρώτη έκθεση αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2017 είχαμε δύο συζητήσεις με οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τελευταία συζήτηση έγινε τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Είχαμε και μία ε, μελέτη που έγινε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ στοχευμένη, που ολοκληρώθηκε τώρα και σύντομα θα δημοσιεύσουμε και τα αποτελέσματα. Πρόκειται για μία έρευνα που προσπαθεί να δει κατά πόσο υποφελούνται από τον σημερινό ορισμό επιχειρήσεις ή όχι. Και επιχειρήσει η οποία θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαΐου. Συγχρόνως έχουμε έναν σύμβουλο ο οποίος αξιολογεί τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ορισμό και το έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί ε, μέχρι το καλοκαίρι. Αν λοιπόν όλα αυτά τα βάλουμε μαζί, θα καταλήξουμε σε κάτι στις αρχές του φθινοπόρου. Ποια είναι τώρα τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μια, θέλουμε να έχουμε έναν ορισμό ο οποίος να επιτρέπει οι επιχειρήσεις που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθεια να μπορούν να υποφεληθούν από αυτήν και όχι άλλε επιχειρήσει οι οποίε υποφελούνται από τα κενά και κάνουν κατάχρηση. Από την άλλη όμω, θέλουμε κάτι απλό που να έχει να κάνει με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, γι' αυτό και πρέπει να είναι απλό. Δεν είναι εύκολο, γιατί μερικέ φορέ αυτά τα δύο είναι αντιφατικά μεταξύ του. Για παράδειγμα, έχουμε δύο κριτήρια σήμερα το δίκτυο κεφαλικής επάρκειας και το προσωπικό. Αλλά για να καθορίσουμε τα νούμερα, από την άλλη μεριά έχουμε και το θέμα της ε, ιδιοκτησίας. Κατά πόσο δηλαδή μια μικρομεσαία επιχείρηση ανήκει σε μια μεγαλύτερη. Ας πούμε αν έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση που δεν έχει άλλους δεσμούς από τη μία, ενώ μπορεί να υπάρχει μια άλλη μικρομεσαία επιχείρηση που αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πώς να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό είναι το περίπλοκο. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Προτείνουμε, όπως λέμε και στην ε, εκτίμηση επιπτώσεων, λέμε τα Πρώτον, να προσαρμόσουμε τα νότατα όρια όσον αφορά το πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Αυτό υπάρχει στις συστάσεις μας. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να καλύψουμε το κενό που έχει να κάνει με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Δηλαδή να εφαρμόσουμε τον ορισμό στις επιχειρήσεις που πραγματικά το χρειάζονται και όχι στις μεγαλύτερες. Και το τρίτο που προτείνουμε στην μελέτη επιπτώσεων είναι να βοηθήσουμε τις νεοφύς επιχειρήσεις που θέλουν να μεγαλώσουν να το κάνουν αυτό παρατείνοντας ίσως ένα-δυο χρόνια την περίοδο αυτή που μεγαλώνει μεν η επιχείρηση, αλλά εξακολουθούμε να τη θεωρούμε μικρομεσαία. Και προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα όσο γίνεται περισσότερο. Διάφορα θέματα έθεσαν ε, οι οργανώσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσπαθούμε να τα λάβουμε υπόψη μας στον ορισμό. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέτει ο εισηγητής σας και οι ευρωβουλευτές. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι το θέμα των mid-caps, της μεσαίας κεφαλοποίησης επιχειρήσεων. Γιατί επαναλαμβάνεται. Εμείς πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα συμπεριληφθούν στον ορισμό των μικρομεσαίων ή θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο χωριστού ορισμού αν συμπεριλάβετε τις mid-caps στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουν να απορροφήσουν την ειδική μεταχείριση πολύ περισσότερο και σε βάρος των μικρομεσαίων. Συνεπώς, ίσως να είναι καλύτερο να υπάρξει διαφορετική πολιτική για τις mid-caps από ό,τι για τις μικρομεσαίες. Το άλλο το οποίο θέσατε είναι τα άλλα κριτήρια, της έντασης εξαγωγών για παράδειγμα ή της κεφαλικής ε, επάρκειας. Και πάλι εδώ το ζήτημα είναι το εξή. Πρέπει να παραμείνουμε απλοί στον ορισμό μας. Και αν έχετε το κριτήριο των εξαγωγών, το είπε κάποιο από τους αξιότιμους ευρωβουλευτές, τι γίνεται με τις παραδοσιακές μικρομεσαίες που δεν εξάγουν, θα αποκλειστούν. Συνεπώ, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και αυτό το στοιχείο. Τι άλλο. Το ζήτημα που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με συστάσεις ή θα έπρεπε να περάσουμε σε μια άλλη νομική βάση, κανονισμό για παράδειγμα. Α, συγγνώμη αν μακρηγορώ. Μη μακρηγορήσετε υπερβολικά, λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, θα ολοκληρώσω σε λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι οι συστάσεις τώρα είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι χώρες ε, μέλη ξεκινούν με μια κοινή βάση και από εκεί και πέρα προσαρμόζονται στις ειδικέ συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα. Ωραία, να ολοκληρώσω εδώ τότε και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, δεν ήθελα να σας ε, σταματήσω στα 20 δευτερόλεπτα. Έχετε δύο λεπτά. Άμα θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε για δύο λεπτά. Όχι, ευχαριστώ. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να απαντήσω, λέει ο πρόσωπος της Επιτροπής. Τώρα, ο εισηγητής. Εμείς ως Επιτροπή Ήτρε είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ήπειρο μας και είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός. Λοιπόν, Μάρκος, μπορείς να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εμπλούτησε ιδιαίτερα η συζήτηση το θέμα και με ενθαρρύνει. Γιατί θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση και τις προτάσεις που γίνονται, είμαστε απόλυτα σε θέση να συμβάλλουμε ουσιοδός σε αυτή τη διαβούλευση. Διότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τα έχουμε το φθινόπωρο. Αλλά τότε είναι αργά για να μπορέσει να συμβάλλει ουσιοδός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να συμφωνήσω με όσους είπαν ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε πολύ τον ορισμό των μικρομεσαίων. Όχι, δεν είναι αυτή η πρόθεση η δική μου. Όχι. Αλλά κοιτάξτε, τα τελευταία 15 χρόνια θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει αλλάξει και μετά από τις ε, ερωτήσεις που κάναμε και στις διάφορες ενώσεις μας είπαν ότι πρέπει να αυξήσουμε κάπως και τον αριθμό των εργαζόμενων και ε, το ύψος του κύκλου εργασιών. Νομίζω ότι αυτή η προσαρμογή είναι μια ιδιαίτερα ε, χρήσιμη προσαρμογή και από αυτού πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε συνένεση. Κάτι άλλο που επανειλημμένα υπόθηκε είναι να μην επικεντρώσουμε ιδιαίτερα στις mid-caps. Αλλά να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτό που μόλις είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ίσως θα χρειαστεί μια ειδική πρόταση για τις mid-caps. Ναι, νομίζω ότι ίσως θα ήταν η καλύτερη λύση. Θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια έτσι. Αλλά, αν δούμε αυτή τη νέα δομή, για παράδειγμα, για τη νέα αμυντική μας βιομηχανία, όλη αυτή τη δομή των διαφόρων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής και που δίνουν τμήματα για κάποια προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερο από 250 ε, εργαζόμενους να έχουν όλα αυτά τα διοικητικά τμήματα. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία. Ε, είστε μια επιχείρηση μέχρι 2.000 εργαζόμενοι, με ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς spin-off έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ένα παράδειγμα που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Ένα άλλο παράδειγμα. Ε, ανησύχησαν ορισμένοι για αυτά που λέμε για τις εξαγωγές. Αλλά γιατί όχι. Εάν επιχειρήσεις ε, ε, εξάγουν ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής τους, έστω και με λίγους εργαζόμενους, γιατί να μην δώσουμε ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτούς. Το ένα είναι ο ορισμός ε, των μικρομεσαίων, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, ιδιαίτερα παραγωγικές mid-caps που θέλουν να αναπτυχθούν, που θέλουν να συμβάλλουν περισσότερο σε κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, γιατί να μην τους δώσουμε νέες δυνατότητες. Αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων πρέπει κάπως να, την, ε, να μπορούμε να την μετρήσουμε, να έχει όρια, να είναι μετρήσιμη. Λοιπόν, όπως είπε και η Κομισιόν, πρέπει να προσαρμόσουμε κάπως κάποιους ορισμούς αλλά επιπλέον πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στις mid-caps με βάση έναν ιδιαίτερο ορισμό. Ε, Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτές ε, τις ε, προτάσεις γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν. Τέλος. Αν θέλουμε να παραταθεί η προθεσμία για τις τροπολογίες μπορούμε να έχουμε δύο εβδομάδες χωρίς ε, να δημιουργήσουμε προβλήματα στο συνολικό χρονοδιάγραμμα. Θα μπορούσα λοιπόν να συμφωνήσω να παραταθεί κατά δύο εβδομάδες. Αλλά σας παρακαλώ να μην επεκτείνουμε τόσο πολύ την ε, ε, προθεσμία, ούτως ώστε να μην προλάβουμε να συμβάλλουμε στις, στη διαβούλευση της Κομισιόν, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκους, για τις παρατηρήσεις σου, λέει ο Πρόεδρος και για την ευελιξία σου. Οπότε, ευχαριστώ όλους όσους ε, παρενέβησαν. Εξαιρετική συζήτηση και από τους Κιώδης ε, και από τους υπόλοιπους και από την Επιτροπή. Μάρκους, θα συμφωνούσαμε λοιπόν ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος έχει περάσει στις 9 Απριλίου Λοιπόν, έχουμε προσθέσει δύο εβδομάδες, όπως πρότειναν κάποιες πολιτικέ ομάδε και συμφώνησε και ο εισηγητή. Οπότε θα μπορούσαμε μάλλον να ψηφίσουμε όπως είχαμε προτείνει και νωρίτερα στις 16 Μαΐου στην Ήτρε και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο τρέχοντος. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Λοιπόν, Να δώσω τώρα το λόγο και την Προεδρία, στην πρώτη Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Πατρίσια, σε ευχαριστώ πολύ για την διαθεσιμότητά σου. Βγάζω την κάρτα μου, βάλει τη δική σου, ωραία, ωραία. Έλα κάτσε εδώ. Ε, άλλαξε και το κουμπί γιατί το έχω γυρισμένο στην πολωνική καμπίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα το αλλάξω λέει η κυρία Τόια. 5 λεπτά διάλειμμα. Γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι τι 10 για να αρχίσει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μπορούμε να αρχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες θα ήθελα να κάνουμε μία δοκιμή πρώτα για να δούμε αν λειτουργούν όλα καλώς. Χαιρόμαστε που είναι ηλιόλουστη μέρα. Όποιος είναι υπέρ του, της ηλιόλουστης μέρας ε, ψηφίζει ναι. Οι υπόλοιποι όχι. Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Τρεις, τρεις, τρεις. Θα ήθελα ο επικεφαλής να το λύσει το θέμα ως προς τους υπεράριθμους. Πλην δύο ακόμα. Παρακαλώ. Ε, βοηθήστε με σας παρακαλώ από το ΕΛΚ. Τέσσερις, τέσσερις ακόμα. Σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Δύο υπεράριθμοι. Scusate, Σας παρακαλώ ε, έχουμε δύο υπεράριθμους και θα ήθελα να ξεκινήσουμε γιατί περιμένουμε εσάς. Ma giusto il sistema, corretto. correct. è corretto. You love this committee too much. Ε, πολύ την αγαπάτε αυτή την επιτροπή. Karis, please. Sorry, you have to resolve this situation. Πρέπει να επιλύσετε αυτό το ζήτημα ε, σε πολύ λίγα λεπτά. Μη χρονοτριβείτε. Karis, please, you have to, to do. Cosa posso fare? Only one more, only one. Ένας υπεράριθμος. Ένας από τους σοσιαλιστές. SD, it's okay. Εντάξει. Υπεράριθμος ένας από το ΕΛΚ. Après, Eh? Madame Viana. Madame? Madame Viana, for the point of Chi è Madame? Madame Viana, S&P. Viana? Sì. No, che nome dice? Madame Viana. Verne, ah. Tu? There's a group, Chairman, if the EPP can't... Εάν δεν μπορεί να λύσει το θέμα το ΕΛΚ, τότε ας μη συμμετάσχει. μέχρι να το λύσει. Mr. Karins, please. This situation is ridiculous. Κύριε Κάριν, σας παρακαλώ. Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το θέμα, γιατί περιμένουν όλοι οι συνάδελφοι. One. Your, please, your, your, please. If your colleagues does it, no, tolga suo. Due. Two. Sorry, I propose that. Two minutes. Δύο λεπτά λοιπόν για να απειλήσουμε το θέμα. Και θα πρέπει να μιλήσουμε το ΕΛΚ. Two minutes. θα ήθελα να αποχωρήσει ο υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Μπορούμε να αρχίσουμε. Ε, Ελπίζω να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις που μαντροπιάζουν. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ. Στην πρώτη μας ψηφοφορία για την οδηγία για το φυσικό αέριο προτείνω μία αναβολή την ψηφοφορία μέχρι να έχουμε τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν. Γιατί με βάση τη Διοργανική Συμφωνία αναφέρεται ότι για κάθε ψηφοφορία χρειαζόμαστε μελέτη αντικτύπου. Παράγραφος 3. Εκεί που λέει ε, εργαλεία για καλύτερη νομοθεσία. Έχουμε ένα αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190. Η ψηφοφορία αυτή δεν προβλέπει συζητήσεις και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο τέσσερις συνάδελφοι υποστηρίζουν τη Μαρτίνα Βέρνα. Πέντε. Εντάξει. Υπάρχει υποστήριξη, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το αίτημα. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ποιος θέλει να αναβληθεί η ψηφοφορία ψηφίζει ναι. So I think you have to make clear ότι πρέπει να διευκρινίζεται πώς θα ψηφίσουμε αν θέλουμε να γίνει τώρα η ψηφοφορία. Ποιος θέλει να αναβληθεί η ψηφοφορία. Αυτοί θα ψηφίσουν ναι. Όσοι δεν θέλουν να αναβληθεί θα ψηφίσουν όχι. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας. Υπέρ ή κατά της αναβολής. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ και πάλι. Εντάξει, ωραία. Πέρας. Το αίτημα αναβολής δεν εγκρίθηκε, άρα θα ψηφίσουμε. Allora, votiamo il rapporto Έκθεση Μπούζεκ. Κοινοί κανόνες, μάλλον, κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά του φυσικού αερίου. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογίες 8, 9, 10, 11 και 12 που θα τις ε, ψηφίσουμε en bloc ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε πάλι έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Ελπίζω να μην πρέπει να το επαναλαμβάνω σε κάθε ψηφοφορία αυτό. Πέρας. Απορρίπτονται. Το αίτημα αυτό απορρίπτεται. Τροπολογία 39, τροπολογίες 39, 35, 36, On block. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 και 6 on block υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται οι συμβαστικές. Τροπολογία 64. 64 και 67 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 68-69 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71, 72, 73 ταυτόσιμες ενία ψηφοφορία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100-101 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστικές 2 και 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137-138 ταυτόσημες υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτονται. 141-142 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Στην αιτιολογική σκέψη 1, το 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 14 και 15 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 με συγχωρείτε ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 16 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία La votazione Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία σε σχέση με το, την εντολή διαπραγμάτευσης, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία και συγχαίρουμε τον κύριο Μπούζεκ, τον εισηγητή.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 Ένας από το έλκα ένας υπεράριθμος πάλι. Εντάξει, πέρας και εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει το 85-86 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Να βγει μια κάρτα παρακαλώ. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές η ε, απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια και πρέπει να ελέγξουμε. 103 ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Προτείνω ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η συμβαστική. 8. Περνάμε στην 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 37. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πρώτον, τελική ψηφοφορία ε, ως προς το τροποποιημένο κείμενο άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση και τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική για την εντολή διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. έχουμε ειδική πλειοψηφία. Ο κύριος Λεβαντόσκι ε, αναλαμβάνει την εντολή, τον οποίο και συγχαίρουμε. Παίρναμε τώρα στην ε, τρίτη και τελική έκθεση. Πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η κυρία Ριβαζή είναι η συγγήτρια. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Προτείνω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται η τροπολογία 21. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Προτείνω ονομαστική ψηφοφορία για να μην χάνουμε χρόνο. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά ως προς τη συμβαστική 8 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. Περνάμε στις επόμενες λοιπόν. 28 με ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όχι ακόμα από ό,τι διαπιστώνω. Πέρας. Εγκρίνεται η 31. 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο, ας γίνει, αν και θα πρέπει να υπάρχει η ίδια, να έχουμε την ίδια πλειοψηφία, άρχεται η ψηφοφορία για την 61. Μία ψήφος ακόμα λείπει πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ας περάσουμε στην ονομαστική για να μην χάνουμε χρόνο. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε την προστίκη στη συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Προστίκη στη συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχετε ψηφίσει ακόμα όλοι. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβαστική 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, με ονομαστική. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Ας γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν ακόμα ψήφοι, δεν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Τροπολογία 59 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας και απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν είναι σίγουρη η κατάσταση. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας και απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, εγκρίνεται λέει η πρόεδρος. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε για την 7 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας και εγκρίνεται σας ευχαριστώ που ζητήσατε επαλήθευση ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψηφίσατε ακόμα όλοι. Πέρας. Η συμβαστική 4 εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και θέλετε να ελέγξουμε την 11. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας και εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη για δεύτερη φορά. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε έναν υπεράριθμο πάλι από το ΕΛΚ. Εντάξει, πέρας και εγκρίνεται. Να συγχαρούμε την συνάδελφο Ριβαζή. Passiamo Πρόεδρε. Όχι, δεν έχει να κάνει μισοφορία για το άλλο θέμα. Γιατί πρέπει να φύγω για το αεροδρόμιο δεν μπόρεσα να βρω το σχέδιο γνωμοδότηση για τι γλώσσε στην ψηφιακή ηλικία στο ίντερνετ και η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι σήμερα. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία αν θεωρούν ότι είναι δημοκρατικέ διαδικασίε αυτέ. Ω κοιόδησε μόλι την προηγούμενη πέμπτη την έλαβα και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ε, βιασύνη γιατί κούλ δεν κάνει τίποτα. Είναι τεχνική ερώτηση. Θα πρέπει να ασχοληθούμε αυτό σήμερα ή όχι.

possiamo continuare. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ. Possiamo continuare allora. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή. Η συνάδελφος Ματίας είναι η συγγήτρια. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε ξέρετε ότι η δυνάμη του άρθρου 54 η Επιτροπή Πολιτισμού είναι η αρμόδια επιτροπή, άρα θα πρέπει και εμείς να συνδράμουμε. Γιατί είναι το ψηφιακό, η έρευνα και άλλες πτυχές που αφορούν τη δική μας επιτροπή. 30 λεπτά η συζήτηση. Το λόγο έχει η εισηγήτρια Ματίας και μετά θα παρέμβουν οι σκιώδεις. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω στο σχόλιο της συναδέλφου σε σχέση με τις πολύ στενές προθεσμίες. Ε, είναι ένα θέμα που δεν μας ικανοποιεί καθόλου, αλλά εξαρτόμαστε από τις προθεσμίες της Επιτροπής Πολιτισμού. Και όπως ξέρετε ήταν ιδιαίτερα μακροχρόνια η διαδικασία για να δούμε εάν υπάρχει επιμερισμός ευθυνών σε σχέση με αυτή την έκθεση μεταξύ κουλτ και ήτρε. Άρα δεν είχαμε αρκετό χρόνο ούτε για τις ε, τροπολογίες, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στα συμπεράσματά μας και δεν κατανοώ αυτό που προαναφέρθηκε σε σχέση με την προθεσμία και τις τροπολογίες. Μίλησα με αρκετούς σκιώδεις ε, ήδη. Τώρα, θα ήθελα να είμαι αρκετά σύντομη, αλλά αυτό το θέμα, όπως ξέρετε, της γλωσσικής ισότητας στην ψηφιακή εποχή είναι η της εποχής. Η πολυγλωσσία είναι το μεγαλύτερο κληροδότημα και η μεγαλύτερη κληρονομιά της ε, Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της ε, ψηφιακής εποχής. Έχουμε 24 ε, επίσημες γλώσσες, έχουμε 60 εθνικές και περιφερειακές γλώσσες και για να υπάρξει χρήση όλων αυτών των γλωσσών χρειαζόμαστε τις κατάλληλες τεχνολογίες, τεχνολογίες εχμής για την διάδοση των πληροφοριών οι γλώσσες αυτές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και θα θέλαμε να δούμε θέματα που άπτονται της δικής μας αρμοδιότητας με βάση την ε, τεχνολογία ή τις τεχνολογίες των γλωσσών για να μπορέσουν να επιβιώσουν όλες οι γλώσσες στην ψηφιακή εποχή θα ασχοληθώ με θέματα που άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων και τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτισμού ήδη συζητήθηκαν χτες. Είναι τέσσερα τα σημεία τα οποία υποβλήθηκαν και εδώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων. Το πρώτο σχετίζεται με τα big data. Ε, ε, ε, όπως γνωρίζουμε, ε, αποτελούν μεγάλο κομμάτι της κληρονομιάς αυτής και θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή πλατφόρμα και στον τομέα της τεχνολογίας καθώς και της τεχνητής ευφυΐας. Αυτό έχει να κάνει και με την έρευνα. Χρειαζόμαστε μία συντονισμένη πρωτοβουλία και ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές γλώσσες και την επάρκεια χρήσης τους, ιδιαίτερα από τα πανεπιστήμια, από τις ΜΜΕ και από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται χρηματοδότηση που θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ε, και στο ένατο πρόγραμμα πλαίσιο και θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μόνο αν έχουμε μία ε, διαλειτουργική πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογική αυτή γλώσσα, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα. Το τρίο το θέμα σχετίζεται με τις ΜΜΕ και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η εργαλειοθήκη που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να γίνονται και πωλήσει, επιγραμμικές ε, πωλήσει προϊόντων και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη και την καινοτομία των ΜΜΕ. Και το τελευταίο σημείο αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν θέλουμε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και εργαζομένων, θα θέλαμε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες στη δική τους γλώσσα. Και γι' αυτό η τεχνολογική επιστήμη των μαζικών δεδομένων θα πρέπει να μας βοηθήσει και να υποβοηθήσει για την καινοτόμα χρήση όλων των γλωσσών. Θα παραμείνω σε αυτά τα τέσσερα σημεία που είναι δικής μας αρμοδιότητας και νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία για να μην ε, εξαλειφθούν οι μικρές γλώσσες οι οποίες έχουν περιορισμένη χρήση στην ψηφιακή εποχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, συναδελφο και περνάμε στους ε, σκιώδεις. Ο κύριος Σαντάργας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Στην εισηγήτρια που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έκανε πολύ καλή δουλειά. Είναι δύσκολο σίγουρα. Η εισηγήτρια κάλυψε το περιεχόμενο, οπότε δεν θα σχολιάσω επί του περιεχομένου. Στηρίζω απόλυτα την γνωμοδότηση αυτή θα ετοιμάσουμε κάποιες τροπολογίες για να υπογραμμίσουμε περισσότερο κάποιες πτυχές της. Όμως θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι έκθεση πρωτοβουλίας, έτσι, γιατί είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει ανάλυση των ευρωπαϊκών γλωσσών και τονίζω ότι εδώ πρόκειται για την πολυγλωσσία, αλλά την τεχνική της πτυχή την τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στα αγγλικά και τις άλλες γλώσσες, τις μεγάλες και τις μικρές, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, τεχνολογικό όμως. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα αυτό καθεαυτό πολυγλωσσίας. Ε, δεν είναι θέμα πολιτισμικό, γι' αυτό και το εξετάζει και η δικιά μας Επιτροπή πολύ σωστά. Τα μέσα για την πολυγλωσία είναι τεχνικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέρετε, ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεράστιες εξελίξεις, αναγνώριση προσώπου κλπ. Αυτές οι εξελίξεις όμως γίνονται και στο γλωσσικό. Ξεπερνιόνται διάφορα προβλήματα, ικανότητες των υπολογιστών κλπ. Ας πάρουμε επίσης το παράδειγμα των αυτοκινήτων με αυτόνομη οδήγηση. Τι σημαίνει αυτό. Αν το αυτοκίνητο μάθει να οδηγάει στα βουνά και μετά το βάλετε στην πόλη με την αυτόμανη αυτή οδήγηση, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική μάθηση. Το ίδιο ισχύει και για το γλωσσικό. Χρειάζονται δεδομένα, big data όπως λέμε, μεγάλα δεδομένα. Και συνήθως στις μεγάλες γλώσσες, στα αγγλικά υπάρχουν, ε, υπάρχει γνώση που θα πρέπει να μεταφραστεί. Άρα είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Η έκθεση αυτή μιλάει και για την μελέτη. Υπάρχει μελέτη που ξεκίνησε από την ΣΤΟΑ και ψάχνουμε για πολιτικές αποφάσεις. ευρωπαϊκή προσέγγιση και λύσεις. προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτήν την ευρωπαϊκή αξία που είναι η πολυγλωσία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Μούντι που αντικαθιστά την κυρία Κούπλα Ευχαριστώ. Πατρίσια. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος, δεν την ακούμε. Ευχαριστώ Πατρίσια. Να ένα παράδειγμα αγγλικών και στηρίζω απόλυτα τα σχόλια των συναδέρφων. Στηρίζουμε λοιπόν την έκθεση αυτή και συμμεριζόμαστε την ανησυχία που λέει ότι πολλές γλώσσες κινδυνεύουν σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Υπάρχει ένα χάσμα που όλο μεγαλώνει ανάμεσα στα αγγλικά και τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες στον τομέα της τεχνολογίας υπάρχουν διαφορετικές ε, περιοχές, χώρες, ε, περιοχές που πλήττονται. Πρέπει η τεχνολογία να είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Τότε θα μειωθεί το χάσμα αυτό. Χρειάζεται και καλό συντονισμό ανάμεσα στην έρευνα και την βιομηχανία. Να προστατεύσουμε τις γλώσσες στον ψηφιακό κόσμο, τις ε, βάσεις δεδομένων και την τεχνολογία να είναι πράγματα διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μείνει μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι. Πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών μελών των πανεπιστημίων και άλλων ε, οργανισμών που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση των γλωσσών. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τα αγγλικά. Σύμφωνα με μελέτη της UNESCO, 35% ε, 50 του περιεχομένου είναι στα αγγλικά. Προκειμένου όμως να εκπαιδεύσουμε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση ολόκληρου του κόσμου, πρέπει να διασφαλίσουμε να υπάρχει μετάφραση των ε, ευρωπαϊκών γλωσσών στα αραβικά, στα κινέζικα ή και ανάποδα. Τα ψηφιακά μέσα που έχουμε στη θέση μας και οι πόροι για τις μικρότερες ε, γλώσσες δεν φτάνει προς το παρόν. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας υπέρ των μικρότερων γλωσσών. Διάφορα προγράμματα τεχνολογίας μετάφρασης έχουν ήδη κατακαιρματιστεί. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει τα πράγματα και να έχει μια εποπτεία του τι ήδη έχει γίνει. Για παράδειγμα μέσω του Horizon 2020, του SP20 κλπ. Θέλουμε επίσης να προσέξουμε τι γίνεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε διάφορα πανεπιστήμια. Για να κυκλοφορήσει περισσότερο η γνώση που υπάρχει ήδη και με μετάφραση των κειμένων, το οποίο θα πρέπει να είναι στο απογελιστικό νέφος. Χρειάζεται επιστημονική γνώση για την μετάφραση και έρευνα. Γι' αυτό κάνουμε έκλειψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει λύσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επιστημονική γνώση θα είναι διαθέσιμη και σε άλλε γλώσσε πέραν των αγγλικών. Φανταστείτε μια κατάσταση όπου επιστημονική γνώση δεν θα υπάρχει για την κλιματική αλλαγή, για το αλκισμό στα φιλανδικά, στα ουγγρικά και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κάτι το οποίο θα πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουν εξίσου πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία και γλωσσικά. Οι τεχνολογίες γλωσσών μπορούν να βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη περισσότερο δίκαια και καλύτερα προσβάσιμη. Ευχαριστώ. Μλιντάρ Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να και τον εισηγητή για την εισηγήτρια δηλαδή για τη θαυμάσια εργασία που βασίζεται στην κατακαιρματισμένη γλωσσική μας ε, πραγματικότητα. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση σε θεσμικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό για την ανάγκη συνδυασμού της πολυπολιτιστικής και πολυγλωσσικής μας ε, πραγματικότητας με τη χορήγηση ισότητας ευκαιριών για τους πολίτες, ε, τους πελάτες και τις επιχειρήσεις για να αξιοποιούν τις ε, τωρινές και μέλουσες εξελίξεις στην ψυχιακή αγορά. Θα πρέπει η ψηφιακή λοιπόν αγορά να μην εξαιρεί κανένα. Αξιοποιώντας ε, τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στην ε, αυξανόμενη ισχύ των υπολογιστών και την επεξεργασία όλο και περισσότερων στοιχείων όπως ε, τα νευροδίκτυα και την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων τεχνολογιών για τις γλώσσες. Και βεβαίως και οι πολίτες πρέπει να έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την πολυγλωσσική δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, δικαιοσύνης, ενέργειας, υγείας και μεταφορών. Η πολυγλωσσία είναι ένα από τα στοιχεία του εμπλουτισμένου ευρωπαϊκού πολιτιστικού μας περιβάλλοντος και αυτό θα πρέπει να δίνει περισσότερες δυνατότητες και στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, γιατί αυτό δεν ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα, πολλοί έχουν προβλήματα και γλωσσικά και τεχνικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα του λιανεμπορίου να αυξήσει το μερίδιό του στην αγορά μέσω επιγραμμικών πωλήσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε οικονομικά την ε, πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω του ε, υπολογιστικού νέφους και όλων των εφαρμογών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες να αξιοποιήσουν την, ε, τις δυνατότητες της αυτόματης μετάφρασης. Θα υποβάλω τις σχετικές τροπολογίες και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιότητες και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τα τέσσερα σημεία στα οποία προαναφέρθηκε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα για να διαχειριστούμε τα μαζικά δεδομένα και έχει μεγάλη σημασία η έρευνα σε αυτόν τον τομέα, τον ε, big data, για να βοηθήσουμε τις ε, ΜΜΕ καθώς και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά στην ουσία τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες πρωτίστως. Και αυτό έχει σχέση και με τους χρήστες ε, του, των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Η πολυγλωσία αφορά μία πολιτιστική κληρονομιά καθώς ε, και μία ταυτότητα, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να ασχοληθεί με την, ε, τις εξελίξεις στον τομέα της χρήσης ε, Gigabyte και να προωθήσει την διαφοροποίηση. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ε, συνεισφέρει αυτή η διαφοροποίηση και η διαφορετικότητα για τη σύγκληση. Οι γλώσσες της ε, τεχνολογίας θα πρέπει να υπηρετήσουν τους πολίτες και γι' αυτό και έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες σε αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία όμως με βρίσκει σύμφωνο. Η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια, θαυμάσια γνωμοδότηση. Η ομάδα μου τη στηρίζει πλήρω. Πολύ σημαντικό ο στόχο μα. Να διασωθούν οι μειονοτικέ γλώσσε ε, από την ψηφιακή εξαφάνιση. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο εάν επενδύσουμε στη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων. Η γνωμοδότηση βοηθάει και θα υποβάλουμε μόνο τροπολογίες για να, προσθέσουμε, να προσθέσουμε ορισμένα επιπλέον στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η τεχνολογία που υπάρχει για τις μειονοτικές γλώσσες εκτός των συνήθων αλφαβήτων ε, πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή πρέπει και οι ε, δημιουργοί λογισμικού και οι κατασκευαστές πληκτρολογίων να κάνουν την αναγκαία προσπάθεια. Και υπάρχει αυτή η στήριξη σε πιο παραδοσιακούς τομείς της ε, κουλτούρας. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον υποτιτλισμό σε μειονοτικές γλώσσες. Θα πρέπει να γίνει άμμος και σε βίντεο και σε άλλες εφαρμογές, γιατί δεν τα παιδιά που μεγαλώνουν με πρώτη γλώσσα, μειονοτική γλώσσα, μπορούν να έχουν τέτοια παιχνίδια μόνο στα αγγλικά ή σε άλλες μόνο μερικές γλώσσες. Άρα δεν μπορούν να μάθουν την μητρική τους γλώσσα, την πρώτη τους γλώσσα αυτά τα παιδιά. Συμφωνώ με την συγκήτρια που λέει ότι είναι σημαντική η χρήση των μεγάλων δεδομένων για να στηριχθεί η ανθρώπινη τεχνολογία. Για παράδειγμα αυτόματη μετάφραση, και επίσης ε, ο τομέας ε, της ε, ηλεκτρονικής γλωσσολογίας πρέπει να ενισχυθεί. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές. Άρα δεν είναι θέμα μόνο ορισμένων εταιριών και ορισμένων ερευνητών και διάφορα προγράμματα στον τομέα της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να στηριχθούν όλες οι γλώσσες για παράδειγμα, ε, ανοιχτή πρόσβαση ε, τεχνολογίε. Είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει να ενισχυθούν. Και να μην ξεχάσουμε και τις γλώσσες ε, για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Τη νοηματική. Τη νοηματική δηλαδή. Δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή γραπτού κειμένου και ε, τα άτομα που έχουν ως πρώτη γλώσσα τη νοηματική θα πρέπει να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Προσβλέπω στη συνεργασία για το θέμα αυτό. Θα είναι πολύ βέβαια σύντομη προθεσμία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ όλων μας και πιστεύω ότι σύμφωνα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πω ότι η Επιτροπή δεν είναι παρούσα και μας είπε ότι θα απαντήσει γραπτό σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Ε, δίνω το λόγο στην κυρία Ματίας και θα ήθελα και εγώ να την συγχαρώ για την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα χρησιμοποιήσω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πολλά από τα θέματα τα οποία έθιξαν και οι υποδείξεις τους είναι ευπρόσδεκτες. Για να συμπληρώσω αυτή την έκθεση, πολλές ε, δεν έχουν συμπεριληφθεί ε, για λόγους χώρου καθαρά, αλλά θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τις τροπολογίες τους γιατί δεν έχω καμία αντίρρηση ως προς αυτές. Θα ήθελα απλώς να πω ότι παρά το γεγονός ότι η λύση δεν είναι η καλύτερη δυνατή, έμαθα από τη γραμματεία ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 12. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, αλλά έχετε λίγο περισσότερο χρόνο για να υποβάλλετε τροπολογίες, οι οποίες όπως σας είπα είναι όλες ευπρόσδεκτες. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ματίας. Έχουμε κερδίσει μία μέρα για τις τροπολογίες. Λίγη προθεσμία αύριο στις 22. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζοντας 2020. Ξέρουμε ότι θα ε, δώσω άμεσα το λόγο στην εισηγήτρια, στην, στην κυρία Ρεμπέκα Χάρμς, αλλά το Συμβούλιο περιμένει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν αποφανθεί ως προς το τελικό κείμενο. Δίνω λοιπόν το λόγο στην ε, Ρεμπέκα Χάρμς για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Καταρχάς ευχαριστώ. Ε, το προσωπικό από την γραμματεία που με βοήθησε και την Κομισιόν. Αλλάξαμε κάπως το χρονοδιάγραμμα εξέτασης της έκθεσης. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά θέματα προς συζήτηση και πρέπει να γίνει προσεκτικά. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά θέματα για την έρευνα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα έρευνας ε, της ε, Ευρατόμ. Μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο και πρέπει. Για μένα δύο ζητήματα πρέπει να τεθούν. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι έχουν αρχίσει να γερνάνε τα πυρηνικά μας εργοστάσια, άρα προκύπτουν πολύ συγκεκριμένα θέματα κινδύνων και ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσουν αυτοί οι κίνδυνοι. Και το δεύτερο, που συζητιέται ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρατόμ, είναι τι θα γίνουν αυτοί οι παγιοί αντιδραστήρες, δηλαδή παροπλισμός, ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων, όχι μόνο των ιδιαίτερα ραδιενεργών καυσίμων, αλλά συνολικά. Η ενδιάμεση αποθήκευση και η τελική αποθήκευση. Αυτό πρέπει να είναι στο κέντρο της έρευνας της Ευρατών. Και αυτό βέβαια πρέπει να απασχολήσει όλα τα κράτη-μέλη, είτε έχουν πρόγραμμα κατάργησης της ατομικής ενέργειας είτε όχι. Η Σουηδία για παράδειγμα πάντα εθεωρεί το, το κράτος μέλος που είχε κάνει τα περισσότερα για την προετοιμασία της τελικής αποθήκευσης. Αλλά πρόσφατα μια δικαστική απόφαση διέκοψε αυτό το πρόγραμμα τελικής αποθήκευσης και οι Σουηδοί θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμά τους για την ε, τελική αποθήκευση ε, θα παραταθεί ιδιαίτερα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο εστίασης της έρευνας αυτό που μου δημιουργεί ερωτηματικά είναι το εξής. Είναι σαφές ότι μειώνεται η χρήση της ε, πυρηνικής ενέργειας στην Ένωση για διάφορους λόγους. Άρα, για ποιο λόγο να αναπτύσσονται και να επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων τύπων αντιδραστήρων και να είναι στο επίκεντρο της ε, έρευνάς μας θα πρέπει να σταθμίσουμε. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την έρευνα για άλλους τομείς παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, πρέπει να αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα όλους αυτούς τους άλλους κλάδους παραγωγής ενέργειας σε σχέση και με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε και που ξέρω ότι το συζητούν και άλλες επιτροπές, για παράδειγμα η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ένας λοιπόν άλλος κλάδος είναι το μέλλον της ε, πυρηνικής σύνδεξης. Μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να έχουμε πραγματικά εφαρμόσιμη έρευνα, ούτε καν να την προσεγγίσουμε. Και έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη κατάσταση από πλευρά χρηματοδότηση ε, αυτή τη έρευνα και πρέπει να συζητήσουμε πόσο θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την έρευνα. Θα πρέπει να γίνει μια ουσιώδη αξιολόγηση και να λάβουμε μια πιο σωστή απόφαση. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τη χρηματοδοτούμε όπω το παρελθόν. Την πυρηνική σύνδεξη πάντα. Αυτά και με χαρά θα ακούσω και πολύ ενδιαφέρον τη γνώμη και των σκιωδών. Ευχαριστώ. Για την παρουσίαση αυτή και το λόγο ε, έχει ο Σκιώδης από το ΕΛΚ. Ο κύριος Σούριτσεκ, ευχαριστώ. Το σημερινό πρόγραμμα Ευρωατόμ προσαρμόστηκε για πέντε χρόνια, 14 μέχρι και 18, στα όρια που θέτει η συνθήκη Ευρατόμ. Όμως η χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια στην έρευνα στα πυρηνικά προβλέπεται ήδη στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Συνεπώς, το θέμα είναι η συνέχιση της έρευνας στα πυρηνικά τα επόμενα δύο χρόνια μετά την εκπνοή του τρέχοντος προγράμματος. Εμείς στηρίζουμε την επέκταση του προγράμματος όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γενικό στόχο την στήριξη της συνέχισης της ασφάλειας όσον αφορά τους τωρινούς αντιδραστήρες και τον παροπλισμό τους. Να λάβουμε υπόψη μας ότι γερνάει ο εξοπλισμός, να φροντίσουμε για πιο μακροπρόθεσμες λύσεις όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα και την τελική τους αποθήκευση, την μεταφορά τους κλπ. Στηρίζουμε επίσης την ε, πραγματογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία προκειμένου και ο κλάδος να φροντίσει για την ασφαλή προμήθεια ε, ραδιενεργών υλικών. Η σύνδεξη επίσης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση. Η χρήση υποδομών έρευνας επίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ των ε, ερευνητών και της γνώσης για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Στηρίζουμε επίσης την ανάπτυξη των κατάλληλων ρητρών ασφαλείας προκειμένου να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την Ευρώπη και παγκοσμίω. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα μέσα στον προτινόμενο προπολογισμό. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις συστάσεις της ομάδας ειδικών της Επιτροπής για άμεσες δράσεις προκειμένου να ενισχυθούν τα αντίστοιχα προγράμματα. Ευχαριστώ. La parola ora al collega le Pellecieri. Engel. Έχει τώρα το λόγο, αλλά δεν είναι. Επειδή δεν είναι παρόν, ο κύριος Μπαλτσίτης έχει το λόγο. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues... Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαμορφώνουμε ακόμα την ε, θέση μας. Οπότε επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω κάποια στοιχεία χωρίς να μπω σε πολλές ε, λεπτομέρειες. Το πρόγραμμα έρευνας Ευρατόμ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία στηρίζουν την απασχόληση και την έρευνα. Και είναι σημαντικό να πετύχουμε τους στόχους μας στον χάρτη πορείας για την σύνδεξη και για άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συζητάμε αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία ε, απομακρύνονται από τα πυρηνικά, αλλά τώρα παγκοσμίως έχουμε περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς από ποτέ. Και πάνω από 40 επιπλέον πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρονικής ενέργειας δημιουργούνται. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα στα πυρηνικά. Αλλιώς θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να έχουμε ε, ηγετικό ρόλο στα πυρηνικά. Δεύτερον, συμφωνούμε με αυτά που λέει το άρθρο 5 για το πρόγραμμα 2020 για τα πυρηνικά που να επεκταθεί σε παραπάνω επικράτειες μετά από την περίοδο 2014-2018 που θα έχουμε το Brexit. Μετά λοιπόν την μεταβατική περίοδο που θα αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρξουν φυσικά αλλαγές και εξελίξεις, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζω και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε τέτοια προγράμματα. Χρειάζεται και συνομιλία με τον κλάδο και μετά το Brexit. Θέλουμε να συμφωνήσουμε για συνεχιζόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την έρευνα και αυτό μακροπρόθεσμα. Προσβλέπουμε σε συνεργασία λοιπόν με την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ρικέτ. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που το Συμβούλιο μας ζήτησε να γνωμοτήσουμε στα πλαίσια αυτής της ε, διαβούλευσης. Πρώτα απ' όλα, από καθαρά δημοσιονομική πλευρά, βλέπουμε ότι αυτή η επανένωση της ε, έρευνας της Ευρατόμ με το ορίζον 2020 και η επέκταση ε, κατά δύο έτη μας επιτρέπει να κάνουμε καλύτερη έρευνα γιατί το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει το εσωτερικό της Ευρατόμ. Δεν έχουμε παρατηρήσει ως προς τα ποσά. Επί της ουσίας. Μπορεί κανείς να έχει διάφορες απόψεις και διάφορες ε, ευαισθησίες για την πυρηνική ενέργεια. Αλλά είναι σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι αιτιολογημένο και πρέπει να υποστηριχθεί. Γιατί σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τα θέματα ασφάλειας των καταστάσεων αλλά και τα θέματα αποβλήτων, αποθήκευσης, λειτουργίας των ε, αντιδραστήρων και γενικά λειτουργίας και αξιολόγηση της λειτουργίας των ε, αντιδραστήρων. Είναι θέμα σε πολλές χώρες, όπως εδώ στο Βέλγιο, αλλά και στις διπλανές χώρες πολλές φορές. Και βεβαίως έχουμε και τις νέες μορφές πυρηνικής ενέργειας, όπου είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα της σύνδεξης. Πρέπει να το στηρίξουμε. Γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, για διάφορα προγράμματα εγγύσεων. Και τώρα βλέπουμε να τίθεται εν κινδύνο. Οπότε μας ικανοποιεί πολύ αυτή η πρόταση που όπως είπε και ο προηγούμενος θα μας επιτρέψει και με τις χώρες που συμμετέχουν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο λόγω των προβλέψεων που γίνεται γι' αυτό θα επιτρέψει λοιπόν και στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει κατά τη μεταβατική περίοδο αποχώρησης. Και ξέρουμε τι σημασία έχει το Ηνωμένο Βασίλειο όχι τόσο πολύ στην έρευνα αλλά στη λειτουργία της πυρηνικής ενέργειας. Η ομάδα μας στηρίζει λοιπόν απόλυτα την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, e. Από την ΚΟΕ e, η Ματίας έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την πρόταση και την εργασία αυτή από τη δική μου πλευρά και στη δική μου ομάδα δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει κοινή θέση ως προς τα ε, πυρηνικά, αλλά μιλήσαμε για την επέκταση του προγράμματος Ευρατόμ και είναι πολύ πιο ευρύ για να το συγχέουμε με την χρήση πυρηνικών. Νομίζω ότι οι πόρους και ανάλογα με τη χρήση θα μπορούσαμε να δεχτούμε αυτή την παρέκταση του προγράμματος. Υπάρχουν ε, βεβαίως αποκλήσεις στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα ε, να πω ότι δέχομαι κατά πολύ αυτά που είπε η εισηγήτρια δεν θα πρέπει ε, να υπάρχει απόκληση αυτού του προγράμματος από το πρόγραμμα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και το πρόγραμμα ενεργειακής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δεν θα πρέπει να προωθήσουμε δράσεις πέρα από αυτές θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή ε, πολιτική αποθήκευσης ραδιενεργού υλικού καθώς και απομάκρυνσης από τα πυρηνικά εκεί που έχει αποφασιστεί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συνέχιση της χρηματοδότησης θα πρέπει να ενισχυθεί και φυσικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία οδό που δεν θα διαιωνίσει τη χρήση των πυρηνικών. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ντεσεβαλιέ από την Ευρώπη των Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζουμε την Ευρατόμ. Καταρχάς, το κείμενο μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην προώθηση της ε, ενέργειας που δεν παράγει οξύδια του άνθρακα, όπως είναι η ε, πυρηνική ενέργεια. Γιατί ορισμένες φορές δημιουργείται εντύπωση ότι μόνο τις ε, ασταθείς μορφές, μορφές ενέργειας προτείνουμε, τις ανανεώσιμες. Η χώρα μου βασίζεται πολύ στην πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν το η Ευρατόμ να μπορέσει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Βρετανούς αν το επιθυμούν ε, τροποδοσία της χώρας τους με σχάσιμα υλικά και για τα, τους αντιδραστήρες ή και για τις ιατρικές εφαρμογές ε, θα συνεχιστεί. Οι Βρετανοί την, πήραν την απόφαση, την κυρίαρχη απόφαση ε, να αποχωρήσουν από την Ένωση. Θα πρέπει να μπορούσαν να αποχωρήσουν χωρίς να κινδυνεύσει η σταθερότητα της χώρας τους. Επίσης, υπάρχει μια ε, συνεργασία και με τους ε, Ρώσους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα μας θεωρεί ότι θα μπορούσε να επεκταθεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την πυρηνική σύνδεξη, που επίση είναι παράδειγμα συνεργασία μεταξύ εθνών για μια μελλοντική ενέργεια που δεν θα παράγει οξύδια του άνθρακα και για μείωση της χρήσης ε, ορυκτών ή καυσίμων. Η Ευρατόμ συνεχίζει να είναι απαραίτητη για τους πολίτες μας. Τα 345 εκατομμύρια που τις δίνουμε ανά έτος είναι μείωση κατά, από την προηγούμενη περίοδο που ήταν 400 εκατομμύρια το χρόνο και μοιάζει περιορισμένη. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά θέματα όπω η ασφάλεια, η ε, διαχείριση των αποβλήτων, την αναφέρατε, και ο παροπλισμός των εγκαταστάσεων και η έρευνα. Μας ικανοποιεί αρκετά το και μου προτείνει η Κομισιόν και ελπίζουμε ο εισηγητή των Πρασίνων να ασχοληθεί, η εισηγήτρια δηλαδή, να ασχοληθεί με το κοινό συμφέρον και όχι με δογματική αντίθεση στην πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Κόλιτσεφ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βέβαια, κανείς μας δεν είναι ειδικό για θέματα πυρηνικής ενέργειας. Είναι πολύ ενδιαφέρον Γιατί πολλές φορές ακούμε ιδεολογικές απόψεις, έτσι, δογματισμούς και όχι απόψεις που να βασίζονται στην τεχνολογία. Θα ήθελα να έχετε υπόψη σας, και να το έχουμε όλοι υπόψη μας, ότι χωρίς την πυρηνική ενέργεια θα αποσταθεροποιηθεί το δίκτυο ε, υψηλού ε, βολτάζου που έχουμε. Άρα ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που αποφασίζουμε τώρα είναι εάν θα υπάρξει και στο μέλλον σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου και αν θέλουμε να υπάρξει εξελεκτρισμός των μεταφορών. Αν τα θέλουμε αυτά χρειαζόμαστε περισσότερους πυρηνικούς αντιδραστήρες, όχι αυτούς μόνο που έχουμε σήμερα. Και το άλλο θέμα που πρέπει να καταλάβουμε. Ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική κατεύθυνση της Ευρατόμ. Αν θέλουμε να συνεχιστεί η, κατάσταση της, η καλή κατάσταση της υγείας μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ιατρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν ραδιοϊσότοπα έχουν πολύ μεγάλη αξία. Πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν η έρευνα και σε αυτό το τομέα. Είναι λοιπόν κατανοητές οι ανησυχίες για τα πυρηνικά απόβλητα, αλλά πολλές φορές ε, είναι δογματικέ αυτές οι αντιρρήσεις. Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι η διάμεση αποθήκευση των αποβλήτων δεν έχει έννοια. Κοιτάξτε, είναι πολύ υψηλής ραδιενέργειας ε, και υψηλής συγκέντρωσης ε, αυτά τα απόβλητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων χωρίς να έχουμε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν για την αιωλική, την ηλιακή ενέργεια. Πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να γίνει έρευνα για την περαιτέρω χρήση ραδιενεργών ουσιών που είναι ήδη διαθέσιμες στην Ένωση. Και τονίζω, θα έχουμε και νέα φάρμακα με ραδιοϊσότοπα τα οποία βοηθάνε πολύ για πολλές ασθένειες. Είναι πολύ πιο δραστικά από τα κλασικά χημικά φάρμακα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και παρακαλώ τους συναδέλφους να τη στηρίξουν και να μην ακούνε διάφορες ε, ε, ε, ε απλοϊκές θεωρίες. Άκρος ενδιαφέροντα όλα αυτά και δίνω το λόγο στη Ρεμπέκα Χάρμς, ε, συγχαίροντάς την και εγώ. Ε, όπως σας προείπα, δεν είναι παρούσα η Επιτροπή, μπορεί να μας δώσει γραπτές απαντήσεις. Η Ρεμπέκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που δεν είναι εδώ η Κομισιόν. Γιατί προκύπτει μια ερώτηση από τη συζήτηση. Ιδιαίτερα από αυτά που είπε ο κύριος Χένκελ η Κομισιόν θα έπρεπε να μας απαντήσει εάν ε, η προσθήκη που έγινε στο άρθρο 5, παράγραφος C, που λέει ότι το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε σύνδεση με χώρες ή περιοχές που ε, συμμετείχαν ως συνδεδεμένες με το 7ο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης 14-18. Εάν λοιπόν αυτή η συμπλήρωση έγινε για να ληφθεί υπόψη το Brexit. Γιατί δεν μου είναι σαφές εμένα. Αλλά είναι θέμα ουσίας. Η Κομισιόν ανήγγειλε ότι θα κάνει μια πρόταση τροπολόγησης της ε, συνθήκης ευρατών, Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα έρευνας που συζητάμε εδώ. Λόγω του Brexit. Λοιπόν, αν δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα την ερώτηση αυτή η Κομισιόν, γιατί ο Γενικός Διευθυντής ε, χάθηκε μεταξύ των κτηρίων της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και δεν μπόρεσε να έρθει μέχρι εδώ, θα πρέπει να μας απαντήσει η Κομισιόν. Θα πρέπει να απαντήσει και στα άλλα θέματα που έθεσε η συζήτηση. Τώρα, για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ίσως να έχουμε διαφορετική πληροφόρηση τώρα για την εξέλιξη της ε, πυρηνικής ενέργειας και στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Μπορώ να σας δώσω πολλά στοιχεία για το πού πάνε τα πράγματα. Μόνο μία χώρα στον κόσμο διευρύνει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Είναι η Κίνα. Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μειώνεται. Αυτό έχει να κάνει για το ότι δεν έχει πια έννοια να υπάρξουν νέοι αντιδραστήρες και έχει να κάνει και με την κατάσταση των μεγάλων επιχειρήσεων του πυρηνικού, όχι μόνο της Αρέβα και της ΕΔΕΦ Αυτές οι δύο είναι περίπου πτωχευμένες. Αλλά και η Westinghouse έχει πτωχεύσει. και έχει επιπτώσεις αυτό συνολικά για τον κλάδο. Και στην Ιαπωνία ο κλάδος μετά τα γεγονότα, την καταστροφή δηλαδή της Φουκουσίμα έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και αυτό είχε λοιπόν παγκόσμιες επιπτώσεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία περαιτέρω επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, όπως είπε ο κύριος Χένκελ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά την ε, πυρηνική σύνδεξη, κάτι πολύ σημαντικό. Γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των ειδικών, την οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς συζητάμε για τον προπολογισμό. Κύριε Χένκελ, μπορεί να γελάτε. Ναι, ναι, όπως γελάτε και για, και για το hashtag MeToo. Ε, αυτά κάνουν ε, ιδίως οι άντρες. Στη συζήτηση λοιπόν για την πυρηνική σύνδεξη μεταξύ των ειδικών υπήρξε μια αλλαγή κατεύθυνσης πέρυσι όσον αφορά την αποτίμηση της ε, αποδοτικότητας της ίδιας της διαδικασίας σύνδεξης. Πόση ενέργεια μπορεί να προκύψει και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Για να δούμε και εμείς ε, πόσο θα χρηματοδοτήσουμε τη σύνδεξη. Νομίζω ότι ο Γέρζι Μπούζεκ συγκάλεσε πολύ πρόσφατα μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που συμπεριέλαβε και τα δημοσιονομικά. Τι θα κάνουμε λοιπόν στο μέλλον, ε, πώς αλλάζει το πλαίσιο, και πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε πόσα θα δώσουμε για τη σύνδεξη. Που από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος του αιώνα δεν θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων ενέργειας που αντιμετωπίζουμε. Αυτή η πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αναγγέλει συναρπαστικό μέλλον για αυτές τις συζητήσεις και νομίζω ότι με βάση τα στοιχεία που θα σας δώσω για την εξέλιξη της, πυρηνικής, της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη και στον κόσμο θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη Ρεμπέκα Χάρμς Τώρα ο Πάτρικ Τσάιντ μόλις κατέφθασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Ρεμπέκα κατά πόσο θα ήθελε να επαναλάβει την πιο σημαντική της ερώτηση γιατί έτσι θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει άμεσα στην ερώτηση. Μπορείς να επαναλάβεις την ερώτηση. Λοιπόν, από τη συζήτηση προέκυψε το θέμα εάν η συμπλήρωση που κάνετε στο άρθρο 5 της πρότασής σας, όπου λέτε ότι το πρόγραμμα Ευρατόμ θα είναι ανοιχτό για τη συμμετοχή συνδεδεμένων, εκεί στο σημείο C, στη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών ή περιοχών που ήταν συνδεδεμένες και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ή το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης 14-18 της Ευρατόμ. Αυτό το βάζετε για να καλύψετε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι καταλάβατε, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη πρώτα απ' όλα που δεν ήμουν εδώ στην αρχή της συζήτησης. Και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ και να συζητήσουμε με την κυρία Χάρμς, ελπίζω κάποια άλλη στιγμή. Πάντω χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Επιτροπή σα την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση τη σημερινή ρύθμιση του κανονισμού Ευρατόμ για την έρευνα και την κατάρτιση. Βασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο της σε μια προσωρινή αξιολόγηση που κάναμε πρόσφατα για το σημερινό πρόγραμμα 2014-2018. Καλύπτει δηλαδή τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών και έμεσες ερευνητικέ δραστηριότητες που είναι από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας με δύο συστατικά που είναι η σύνδεξη και η σχάση. Περιορίζει η συνθήκη βέβαια την περίοδο στα πέντε χρόνια. Και γι' αυτό και υπάρχει διαφορά όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό για την έρευνα και την κατάρτιση, το πρόγραμμα αυτό Ευρατόμ δηλαδή. Μας εθαρρύνουν πάντως τα αποτελέσματα της προσωρινής αξιολόγησης, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι γενικά μιλώντας το πρόγραμμα λειτουργεί καλά, ικανοποιητικά και ιδιαίτερα μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα στο, στην Ιαπωνία πριν από πέντε χρόνια, όπως γνωρίζει η Επιτροπή σας, οι έρευνες σε θέματα πυρηνικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνονται κυρίως στην πρόληψη, μάλλον αποκλειστικά στην πρόληψη. Ασφάλεια, προστασία, ε, διασφάλιση και ακριβώς ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι πράγματι και τα κράτη-μέλη εκεί πρέπει να βάλουν ε, το κέντρο βάρους. Συνεπώς, συντάσσοντας την πρότασή μας για την επέκταση της περίοδου και το 2019 και το 2020, συνεχίζουμε με το κείμενο, η κύρια αλλαγή είναι αλλαγή στα νούμερα του προπολογισμού. Αλλαγή που απορρέει από τη συμφωνία στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι πρώτες συζητήσεις με τις χώρες μέλη στο Συμβούλιο ήταν αρκετά παραγωγικές, προχωράμε καλά και επιβεβαιώνουν ότι η βάση και των προηγούμενων προγραμμάτων θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και αυτήν την επέκταση τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι όντως πρέπει να γίνει. Βέβαια περιμένουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να απαντήσω για τις συνδεδεμένες χώρες. Η διάταξη στην οποία αναφέρθηκαν οι ευρωβουλευτές δεν πρόκειται ρητά να αναφέρει την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή σα, γίνονται συζητήσεις για τις μελλοντικέ σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάντως, αν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων λένε ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή του προγράμματος, τότε θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Πάντως οι διατάξεις στο κείμενο ως έχουν τώρα μιλούν για άλλες δεδεμένες χώρες που ήδη έχουν σχέση συνδεδεμένου κράτους με την Ευρατόμ. Είτε με το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατόμ, είτε με το πρόγραμμα καινοτομίας και έρευνας 2014-2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έληξαν οι πρωινές εργασίες και πολύ νωρίτερα από το προσδοκόμενο. Έχουμε μία ώρα επιπλέον στη διάθεσή μας και θα τα πούμε στις 2.30 με την εισηγήτρια Βιόλα για το